επί τη ευκαιρία τη παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων τη Προεδρία τη Ρουμανίας και επί τη ευκαιρία θέλω να καλωσορίσω την Πρωθυπουργό της Ρουμανικής ε, Δημοκρατίας, την παλαιά συνάδελφο κυρία Νταντσίλα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας ως Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Ανέλαβα την εντολή της Προεδρίας από την Αυστρία και θα ήθελα να πω με αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ μάλλον στις ευχαριστίες μου προς την Αυστριακή Προεδρία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Φιλανδία και την Κροατία γιατί είχαμε μία πολύ καλή συντονιστική δραστηριότητα για ένα κοινό πρόγραμμα για τους επόμενους 18 μήνες. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη ήξερε από πάντα να ξεπεράσει προς κόμματα και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βασίστηκε στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Σήμερα Βρισκόμαστε εκ νέου στη πολλωστή διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Όπως ξέρετε, κάθε τέτοια κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και νέα αρχή. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα με το δικό μας όραμα για τους επόμενους έξι μήνες ε, δεν ε, μιλάμε απλούστατα για μία επίσημη εντολή. Έχουμε 500 εκατομμύρια που αναμένουν απάντηση από την Ευρώπη. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εργάζονται για τους πολίτες και φτάνουν σε αποτελέσματα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Γνωρίζω ότι το πρώτο στάδιο της εκπεριτροπής προεδρίας θα, είναι, θα αποτελείται από εντατική εργασία σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη για να ολοκληρώσουμε πολλά θέματα που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε προκλήσεις. Το δικό μας πρόγραμμα βασίζεται στην συνοχή ως κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις, τις διαστάσεις πολιτική, έτσι ώστε να υπάρχει ένωση μεταξύ κρατών μελών, οικονομική και εδαφική συνοχή και μείωση των πολλαπλών ταχυτήτων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών, καθώς και κοινωνική συνοχή για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις τέσσερις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η πρόσληψη πραγμάτων θα πρέπει να ακολουθήσει μία εγκάρσια πορεία με βάση τις θεματικές μας και με βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες, δηλαδή Ευρώπη της σύγκλησης, της ασφάλειας, της Ευρώπης των κοινών αξιών και του παγκόσμιου παράγοντα. Η Ευρώπη της σύγκλησης είναι ο πρώτος πυλώνας δράσης της Ρουμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο για την διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ανέλυξης και μείωση ανισοτήτων, ανταγωνιστικότητα και συνδεσιμότητα, καθώς και ένωση των αγορών. Αυτός είναι ο πυρήνας της, οικονομικής, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ένας από τους στόχους της Ρουμανικής Προεδρίας είναι να προωθήσει τα νομοθετικά ζητήματα μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς για να έχουμε μία χρηστή λειτουργία της αγοράς. Θα πρέπει να παγιοποιήσουμε την επιστημονική και τεχνολογική βάση των βιομηχανιών έτσι ώστε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο και μπορούμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας. Αυτό αφορά και την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ψηφιακή επίθεση έχει προωθηθεί ήδη και από τους Εσθονούς και τους Αυστριακούς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπό τον ίδιο ρυθμό. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη λειτουργική διασύνδεση Ανατολής Δύσης, Βορρά και Νότου για να προωθήσουμε αυτές τις τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας, οικονομικής ανταγωνιστικότητας και προώθησης των πλέον απομακρυσμένων περιφερειών. Θέλουμε μία νέα πολιτική στον βιομηχανικό τομέα, αλλά έχει μεγάλη σημασία και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς. Αυτά τα θέματα κατέχουν έχουν σημαντική θέση στην Προεδρία μας. Ο δεύτερος πυλώνας της Ρουμανικής Προεδρίας αφορά την Ευρώπη της ασφάλειας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που απειλούν τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και απειλών που υποσκάπτουν την ευημερία της ανοιχτής μας κοινωνίας σε έναν κόσμο επιταχυμένη σε ψηφιοποίηση θα πρέπει να προωθήσουμε την προστασία των πολιτών στον εικονικό κόσμο. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε την ανθεκτικότητα της Ένωσης ως προς τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία για οποιοδήποτε πρόγραμμα που αφορά τον τομέα της ε, πληροφορικής. Στο πλαίσιο της ασφάλειας θα προωθήσουμε και τις διαπραγματεύσεις μας και τις πρωτοβουλίες για να έχουμε μία συνεκτική προσέγγιση των ροών της ε, μετανάστευσης, την ενδυνάμωση των συνόρων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προώθηση της ασφάλειας των πολιτών στον εικονικό κόσμο, καθώς και επέκταση της εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Επίσης, συνεργασία της δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστικών αρχών στο θέμα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Θα θέλαμε λοιπόν να προωθήσουμε τη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες ε, διαμετακόμισης στα πλαίσια των μεταναστευτικών ροών. Το τρίτο θέμα είναι η Ευρώπη ως παγκόσμιος ε, δράστης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κοινέ ε, αποφάσεις όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας θα θέλαμε να ενισχύσουμε την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια ενός συμπληρωματικού χαρακτήρα δράσης ως προς το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σχέσεις άμεσης γειτονίας για να προωθήσουμε τις δράσεις μας. Δέκα χρόνια μετά τις δέκα χρόνια μετά την απαρχή των εταιρικών σχέσεων με τις ανατολικές χώρες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια. να δούμε και ποια θα είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκακέρα. Να εξυγχρονίσουμε το πολυμερές εμπορικό πλαίσιο καθώς και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις σε διεθνές επίπεδο. Μιλάμε για μια Ευρώπη κοινών αξιών. Για να προωθήσουμε λοιπόν την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίσει η κοινωνία μας όπως ο ε, ρατσισμός, μυσαλλοδοξία, ξενοφοβία, αντισημιτισμός και ρητορική μίσους θέλουμε μία πιο δημοκρατική κοινωνία, γι' αυτό θα μιλήσουμε για ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων, όπως επιθυμούν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για την αξιοπιστία μας εναντί των πολιτών. Αυτό το λέω και από την πλευρά της Ρουμανίας, την οποία εκπροσωπώ και ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει μια άνηση μεταχείριση της ε, Ρουμανίας τη στιγμή που επικρίνεται η χώρα μας για θέματα τα οποία γίνονται ανεκτά όσον αφορά άλλα κράτη-μέλη. Και για τη Ρουμανία υπάρχουν συγκεκριμένες ε, ρήτρες αιρεσιμότητας που δεν ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη. Επίσης παραμένουμε εκτός χώρου Σέγγεν και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ζαν Κλόντ Juncker και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη γιατί μας υποστήριξαν για την προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Αυτά όλα τα αναφέρω για να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένες ευρωπαϊκές αποφάσεις συρρυκνώνουν το πλαίσιο δράσης συγκεκριμένων πολιτών και μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους πολίτες των κρατών μελών που εμπλέκονται και δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση πολιτών κρατών μελών. Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν το κλειδί δράσης μας σε ατομικό επίπεδο και συλλογικό μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινή μας δραστηριότητας. Θα πρέπει οι νέοι να συμμετέχουν στη διαδικασία οικοδόμησης μιας δυνατής Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε τις αποφάσεις ε, του Βρετανικού Κοινοβουλίου ως προς το Brexit και είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει άμεσα τη Ρουμανική Προεδρία. Θα λάβουμε λοιπόν υπόψη τα νέα αυτά δεδομένα και θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την κατάσταση. Το Μάιο Επίσης θα εκλεγεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να λάβουμε υπόψη αυτή τη νέα εκλογική διαδικασία γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε μία πιο δυνατή Ευρώπη με βάση τις ιδρυτικές ε, αξίες της και με βάση τις ευρωπαϊκές γενικότερα αξίες. Πιστεύω σε μια Ευρώπη μέσω της ενότητας, μέσα στα πλαίσια της τήρησης των εντολών και καθηκόντων και πιστεύω σε μια πιο ευρωπαϊκή Ευρώπη μέσα στα πλαίσια των κοινών αξιών και τη συμμετοχή των πολιτών που θα πρέπει να νιώθουν ότι ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο μία ενωτική Ευρώπη, μία ενωμένη Ευρώπη στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα που αποτελεί μία πολύ καλύτερη λύση για όλα τα μελλοντικά μας προβλήματα και την αντιμετώπιση τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπρόεδρος της το Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντα εκ μέρου του Πρόεδρου Γιουνκέρ, εκφράζω την χαρά και ικανοποίησή μου που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την πρώτη στην ιστορία Ρουμανική Προεδρία. Η Ρουμανία, όπως και η Εστονία, η πατρίδα μου, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, γιόρτασαν την εκατοστή του επέτειο πέρσι επέτειο από την ίδρυση. Στιγμή σημαντική για να κοιτάξουμε και προς, το, προς τα πίσω, να δούμε τι έδαφος έχουμε διανύμησει σε αυτά τα χρόνια. Η Ρουμανία έχει διανύσει σημαντικό έδαφος λοιπόν και βρίσκεται τώρα στη θέση που της ανήκει, στο κέντρο της Ευρώπης. Καλύτερο σύμβολο αυτής της προόδου δεν μπορούσε να είναι άλλο από την Προεδρία αυτή στο επόμενο εξάμεινο η Ρουμανία θα ηγηθεί του Συμβουλίου των Υπουργών σε μια κέρια σημασία εποχή για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι με τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό τη, όπου παρακολουθήσαμε και το πολύ καλό επίπεδο των προετοιμασιών, αλλά και τον ενθουσιασμό που εμπνέει την κυβέρνηση για το έργο που έχει μπροστά της. Προεδρία όμως σημαίνει ταυτόχρονα και ευθύνε πάνω απ' όλα σε περίοδους ε, αλλαγών, εξελίξεων και προεκλογικών εκστρατιών. Όπως πολλές φορές έχει επισημάνει ο πρόεδρος Γιονκέρ, η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας. Είναι έτοιμη να σας στηρίξει σε κάθε βήμα της πορείας σας. Θα εργαστούμε χέρι με χέρι με όλα τα θεσμικά όργανα, με όλους τους θεσμούς και τις, ε, τους αρμοδίους που θα εμπλακούν σε αυτήν την ε, Προεδρία για το επόμενο εξάμεινο σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης. Μπορείτε να υπολογίσετε λοιπόν σε εμά. Όπω όμω υπολογίζετε εσεί σε εμά, μπορούμε και εμεί να υπολογίζουμε σε εσά. Υπολογίζουμε στο ηγετικό σα πνεύμα, τη σταθερότητά σα, την ικανότητά σα να χτίσετε γέφυρε, να οικοδομήσετε συνένεση τόσο στην Ευρώπη όσο και στα εσωτερικά σα. Και αυτό το λέω γιατί κάθε επιτυχημένη Προεδρία πρωταρχικά και πάνω απ' όλα εξαρτάται από την εθνική ενότητα και την πολιτική συνένεση. Ένα ενωμένο μέτωπο λοιπόν στο εσωτερικό της χώρας θα βοηθήσει να προχωρήσει μια ενωμένη Ευρώπη. Η Ρουμανία γνωρίζει καλύτερα από πολλές άλλες χώρες το δύναμη της ενότητας. Κατά την προετοιμασία για την ένταξη στην Ένωση στάθηκε ολόκληρη η χώρα ενωμένη και εργάστηκε για να εξασφαλίσει πως θα εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια προσχώρησης. Η επιχείρηση αυτή, η προσπάθεια αυτή δεν ήταν απλώς μία ε, επιβεβαίωση σε κουτάκια των ε, προϋποθέσεων που πρέπει να πληρωθούν. Ήταν η προετοιμασία για ένταξη σε μια ένωση κοινών αξιών, ελευθερίας, δημοκρατίας, κράτους δικαίου, αυτών των αξιών για τις οποίες αγωνίστηκε η χώρα, αυτών των αξιών που ποτέ δεν μπορούν να ε, μειωθούν ή να αποδυναμωθούν. Το επόμενο εξάμεινο, αλλά και πέρα από αυτό, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Αξιότιμοι βουλευτές, άρχισα την ομιλία μου λέγοντας ότι κάθε Προεδρία συνοδεύεται από ευθύνη για όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό θα είναι το καθήκον της Ρουμανίας στο επόμενο εξάμεινο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο στο μέλλον. 242 προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν κατατεθεί πρέπει να εγκριθούν από τους συνομοθέτες. Θα είναι πολύ περιορισμένο το διάστημα αυτό που θα έχετε στη θέση σας για να καλύψετε αυτά τα καθήκοντα καθώς το Κοινοβούλιο 18 Απριλίου σταματάει τις εργασίες του για να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Αυτές οι 242 ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεγαλύτερο τους ε, τμήμα αφορούν πάρα πολύ σημαντικά κέρια για την Ευρώπη θέματα όπως ε, το Brexit, η μετανάστευση και άλλα. Ο δικός μου τομέας της ψηφιακής οικονομίας έχει περίπου 30 προτάσεις που πρέπει ακόμη να εγκριθούν. και αφορά πάνω απ' όλα προτάσεις που θα φέρουν σημαντικές αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή του Ευρωπαίου. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει, κάνει κανείς αγορές πέραν των συνόρων ηλεκτρονικά το δικαίωμα στην προστασία της προσωπικής ζωής στο διαδίκτυο, της προστασίας από τις κυβερνοεπιθέσεις, περιλαμβάνεται σε αυτές τις προτάσεις. Εταιρικοί κανόνες ε, που έχουν τα χαρακτηριστικά των κανόνων του 21ου αιώνα. Κανόνες για τον ψηφιακό κόσμο σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για τον προσοχή προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ δεν μιλούμε για αριθμού ή για δεκαδικά ψηφία. Εδώ μιλούμε για αποφάσει που θα κρίνουν το μέλλον τη Ευρώπη, θα ορίσουν το τι είδου Ευρώπη θέλουμε για το μέλλον. Είναι το μέλλον μα, εκφρασμένο σε αριθμητικού όρου. Γιατί ο προπολογισμό θα δείξει στον Ευρωπαίο ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να πάρει στα χέρια τη το μέλλον της. Όταν ε, συνέλθουν στο Συμπίου στις 9 Μαΐου οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να είμαστε θέση να δείξουμε πως έχουμε προοπτική για μέλλον, για ένα μέλλον πιο ισχυρό, πιο ενωμένο, ένα, ένα μέλλον μιας Ευρώπης με ηγετική θέση και ενωμένης. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα πάρει μαζί του Ευρωπαίου όταν προσέλθει στην κάλπη λίγες μόνο εβδομάδες αργότερα ιδιαίτερα για αυτούς που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν, θα έχει κρίσιμη σημασία. Είτε πρόκειται για ψηφοφόρους των κρατών της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά ή του Νότου της Ευρώπης, όλοι αυτοί οι νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θέλουν ένα μέλλον πιο φωτεινό, πιο αισιόδοξο. Θέλουν μια Ευρώπη ενωμένη, που θα αναπνέει με τους δύο τις πνεύμονες, και τον Ανατολικό και το Δυτικό, που θα ενώνει όλες τις πλευρές της Ευρώπης. Πρέπει να τίνουμε λοιπόν χειρά βοηθεία σε αυτούς τους νέους, να τους δώσουμε το χέρι και να τους δείξουμε ότι η Ευρώπη αναπτύσσεται για το δικό τους καλό. Και αυτό είναι το καθήκον που έχει να επιτελέσει η τρέχουσα Προεδρία της Ρουμανίας. Γι' αυτό θέμασε στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουμε να το υλοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μουτσομέσικα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Στόλογιαν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλωσορίσατε κυρία Πρωθυπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πρόεδροι των ε, θεσμικών οργάνων σας υποστήριξαν, εξέφρασαν την υποστήριξή τους εκ των προτέρων της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Μετανάστευση, κινητοποίηση στις μεταφορές και περίπου 40 εκθέσεις που αφορούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 και από τις λύσεις που θα δοθούν, οι λύσεις μάλλον που θα δοθούν, θα αποτελέσουν πρόκριμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πορείες της. Έχετε πολλούς νέους υπουργούς που δεν έχουν πείρα στις διαπραγματεύσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσετε από αυτούς τους υπουργούς να βασίζονται στις ε, συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της μόνιμης ρουμανικής αντιπροσωπείας που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα αυτά. Μιλήσατε πολύ σωστά για την ανησυχία που υπάρχει ως προς τις ε, πρώην ανατολικές χώρες που δεν θα πρέπει να μείνουν στο απόκεντρο της ένισης. Αλλά, όπως ξέρετε, η Ρουμανία δεν ανήκει ούτε στην Ευρωζώνη ούτε στο χώρο Σέγγεν. Άρα είναι πλήρες μέλος, αλλά με σοβαρές ελλείψεις. Οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τόνισαν ότι θα υποστηρίξουν τη Ρουμανία στην προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Όμως, ως Πρωθυπουργό έχετε υποχρεώσεις έναντι όλων των πολιτών της Ρουμανίας και του επιχειρηματικού χώρου να συναντηθείτε με τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας και της Γαλλίας, με τους καγκελάριους της Αυστρίας και της Γερμανίας και να τους πείσετε ότι η Ρουμανία είναι έτοιμη να προσχωρήσει στο χώρο του Σέγγεν. Στην Ολλανδία θα πρέπει να μεταβείτε και στη Βουλή των Κοινοτήτων και επίσης δεν υπάρχει αξιοπιστία τη, όπως ξέρετε, του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα της Γερουσίας. Ως προς την Ευρωζώνη, μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας προσχώρησης, είπατε ότι θα δημοσιοποιήσετε το πρόγραμμα δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2018 παρήλθε και δεν έχουμε ακόμα αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα να επιταχύνετε τους ρυθμούς σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην άσκηση της Ρουμανικής Προεδρίας. Εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Ούντο Μπούλμαν έχει το λόγο. Αγαπητή Πρωθυπουργέ, αγαπητή Βιορίκα, καλώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγχαρητήρια επί τη ευκαιρία της ε, ανάληψης ε, της Προεδρίας από τη Ρουμανία. Όλοι γνωρίζουμε την προσωπική σας ε, αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πρώην συνάδελφο σας γνωρίσαμε ως πάρα πολύ στρατευμένη Ευρωπαία και πραγματικά αυτό αποτελεί τη βάση για μια αγαστή συνεργασία μας με τη Ρουμανική Προεδρία δεδομένων και των όσων μας περιμένουν που τα αναφέρατε και της σοβαρής κατάστασης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Άκουσα την ομιλία σας με ενδιαφέρον και έχετε δίκιο. Η περιφερειακή συνοχή, η κοινωνική συνοχή είναι ένα θέμα αποφασιστικό και εγκάρσιο. και αυτή η ιδέα να οργανώσουμε με νέο τρόπο την ευρωπαϊκή σύγκληση θα πρέπει να κυριαρχεί στις συζητήσεις μας. Οι τελευταίες ώρες σήμερα έδειξαν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Λονδίνο και πόσο ακόμα έργο απομένει να γίνει μέχρι την ε, απόφαση απόψε θέματα φορολογικά, θέματα χρηματαγορών θα πρέπει να μας απασχολήσουν, να τα ε, επανακαθορίσουμε και το μεταναστευτικό είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα. Θα ήθελα εδώ να σας επενέσω και να αποτίσω ένα φόρο τιμής σας, γιατί κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αποφασίσατε να ενταχθείτε στο στρατόπεδο εκείνων που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στη Μεσόγειο, να σώζουν ζωές και όχι να εθελοτυφλούν απέναντι στα όσα συμβαίνουν ή να ενταχθούν στη λέσχη εκείνων που ήδη πανηγυρίζουν για την ε, διαφορία τους. Ε, θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε προβλήματα που έχουμε και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μας ανησυχούν. Πολλά ε, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα ε, στη Ρουμανία. Θα πρέπει να παταχθεί, να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά. Αν στην Ευρώπη υπάρχει τέτοια κατάσταση να ε, επηρεάζουν οι μυστικές υπηρεσίες τη δικαιοσύνη και την εισαγγελία. Αυτό είναι απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι. Το αναφέρω εδώ, αλλά θα πρέπει να το συζητήσω και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ε, της Ρουμανίας, γιατί στη δική του αρμοδιότητα είναι μυστικές υπηρεσίες. Οπότε, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλή ε, ομόνια, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και να αποδίνουμε και τις ευθύνες εκεί που ανήκουν. Τώρα θα μιλήσω για, πράγματα ε, τα οποία ορισμένοι λένε πίσω από την πλάτη κάποιον. Εγώ όμω τα λέω ξεκάθαρα εδώ. Αν στη χώρα σα υπάρχουν αδικίες από τη δικαιοσύνη, ε, θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι η απάντηση γενική αμνηστία, γιατί βάζει δίκιο και άδικο στο ίδιο τσουβάλι. Θα πρέπει να ε, κυριαρχήσει το κράτο δικαίου εκεί που χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Γνωρίζω ότι το επιθυμείτε και θέλω να σα ενθαρρύνω. Κάντε το αυτό γιατί ε, αυτό θα διευκολύνει και την Προεδρία σας και σας προσωπικά και τη χώρα σας και θα έχετε την Ευρώπη στο στο αν το κάνετε. Το κράτος δικαίου είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών που προστατεύει τους ανθρώπους, εγγυάται τις ελευθερίες απέναντι στο κράτος και τερματίζει την αυθαίρετη κυριαρχία. Αυτό ισχύει έναντι όλων. Τα γνωρίζουμε εμείς αυτά οι σοσιαλδημοκράτες, γιατί 150 χρόνια αυτό ε, υπερασπιζόμαστε παντού όπου κινδυνεύει. Αλλά ε, το κράτος δικαίου ε, δεν ε, μπορεί να χρησιμοποιείται ε, ως πρόφαση και πρόσχημα από τους πολιτικούς αντιπάλους για να γίνουν κάποια πολιτικά παιχνίδια. Κυρία Πρωθυπουργέ, εσείς είστε μια γυναίκα θαραλέα και το γνωρίζω. Η μεταρρύθμισή σας μπορεί να αποτελέσει θαυμάσια προϋπόθεση για τη συνεργασία μας στο επόμενο εξάμεινο. Και να πω κάτι σε κάποιους παντογνώστες εδώ, ιδιαίτερα ε, τους ανταγωνιστές σας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αν αυτές τις μέρες υπάρχει μια χώρα που κλείνουν πάλι πανεπιστήμια, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ από το φασισμό, ε, ε, που υπονομεύονται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και φημώνεται ο κόσμος, τότε να πάτε να τα πείτε και στον κύριο Όρμπαν, γιατί δεν τολμάτε να το τα πείτε κατάμουτρα δεν χρειάζεται να σκουπίζετε τα παπούτσια σας στην ε, επερχόμενη Προεδρία. Είναι λάθος αυτή η κατάσταση. Η Ουγγαρία είναι το πρόβλημα. Τα είχα πει και στον κύριο Γιούγκερ προσωπικά. Έτσι θα, θέλω να τα λέμε και αυτά εδώ. Εκ μέρου των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, κυρία Στίφενς. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρωθυπουργέ, καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά και να καλωσορίσω και τη Ρουμανική Προεδρία. Έξι μήνε είναι μια σύντομη περίοδο για να συζητήσει κανεί και να διαπραγματευτεί. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να συντονιστούμε μαζί με τι δύο επόμενε Προεδρίε. Για τη Ρουμανική Προεδρία, η ευρωπαϊκή διεύρυνση είναι ήδη μια προτεραιότητα για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2018 εκφράζει την φιλοδοξία να διευρυνθεί. Αν κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, μπορούν έξι χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια να έχουν ενταχθεί περί το 2025. Καλύτερα όμως θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει κατά, ε, τάξη ε, στα εσωτερικά της και σας παραπέμπω στο Brexit, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών ε, για το μεταναστευτικό και την ε, πολιτική μας. Για μας αυτή είναι η προτεραιότητα, η λάθρομετανάστευση και ε, παρακαλώ να ακολουθήσουμε το αυστραλιανό μοντέλο ε, που αποθαρρύνει τις παράνομες αφήξεις. Ελπίζω να συμφωνήσετε και να το συζητήσετε αυτό στις διαπραγματεύσεις ε, όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί το κοινοτικό κεκτημένο για το άσυλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Άλντε, ο κύριος Φερχόφστατ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ. Η χώρα σας αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια θα έλεγα πολύ κρίσιμη στιγμή αμέσω πριν τις ευρωεκλογέ. Έχω ετοιμάσει ένα κατάλογο πακέτο κινητικότητας και μεταφορών, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που χρειάζεται συμφωνία και βεβαίως πολύ σημαντικό δύο διαδικασίες άρθρο 7 μία κατά της κυβέρνησης της ε, Πολωνίας και μία που έχει ε, θέσει σε κίνηση το Κοινοβούλιο κατά της κυβέρνησης Ορμπάν. Πολύ δουλειά λοιπόν έχετε μπροστά σας και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί, να έχουμε και τρίτη περίπτωση άρθρου 7 κατά της ρουμανικής κυβέρνησης αυτή τη φορά. Γιατί θα σας το πω, έχω την εντύπωση πως δεν απέχετε πολύ από αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή καθώς συνεχίζεται να αγνοείται τις ε, γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας και για ορισμένα νομοθετικά ε, κείμενα, νομοθετικές προτάσεις που έχει ενώπιόν του το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο της Βουλής και επικεφαλής του κόμματος, τον κύριο Τρεκνέο, ο οποίος της τάσης της πλειοψηφίας σα είπε «Α, το κράτος δικαίου είναι θέμα ε, επικουρικότητας». Όχι, ένα λεπτό. Επικουρικότητα μπορεί να είναι για πολλά θέματα ισχυρός κανόνας, αλλά όχι για το κράτος δικαίου. Δεν εμπίπτει στην επικουρικότητα το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς το ίδιο, την ίδια ακριβώς μέρα, είπα και στον κύριο Ντεριτσάνου, ο οποίος μου έδωσε την υπόσχεση πως η κυβέρνησή σας και τα δύο κόμματα που σχηματίζουν την κυβέρνηση συνασπισμού θα δεχθούν τις προτάσεις αυτές και θα συμμορφωθούν απολύτως στις νομοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Πολλοδεμάλλον συμφώνησε μαζί μου πως η Επιτροπή της Βενετίας θα κληθεί να ε, εκφέρει δεύτερη γνώμη άπαξ δηλαδή και οι προτάσεις αυτές προσαρμοστούν, θα αποσταλούν και πάλι στην Επιτροπή της Βενετίας Και πρόκειται για προτάσει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, για τον ποινικό κώδικα, για την ε, ποινική δικονομία και για την νομοθεσία τη σχετική με τις μη κυβερνητικέ οργανώσει. Θα πρέπει να σας επισημανώ με απόλυτη ειλικρίνεια πως από την ε, συνάντησή μας εκείνη που ήταν και ο κύριος Μπούλμαν και άλλοι στο, Βουκαρέ, στο καμία από τις ε, υποσχέσεις αυτές είναι δεμένα, υλοποιούνται. Η χώρα, η κυβέρνηση σας συνεχίζει στο δρόμο των χείριστων πρακτικών των άλλων, όπως του Ορμπάν και του Κασίνσκι. Και επιπλέον, σας ερωτώ, αληθεύει αυτό που διαβάζω στον τύπο, ότι δηλαδή σκοπεύετε να υιοθετήσετε νόμο που θα, χορηγήσει, θα χορηγεί αμνηστία για τις περιπτώσεις διαφθοράς δηλαδή οι μεγαλοκαρχαριές θα είναι εκτός του ελέγχου των δικαστηρίων. Ένα πολύ απλό πράγμα θα σας πω με την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η δική μου η πολιτική ομάδα και η πολιτική οικογένεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει το δρόμο της ε, συνένεσης και δεν θα σας αφήσει ήσυχος. Θα θέλουμε να σταματήσει αυτή η πορεία. Θέλουμε να καθαρίσει η χώρα από τη διαφθορά και την κατάχρηση της εξουσίας από την παλαιά μυστική υπηρεσία. Και αυτό δεν αποτελεί επίκριση για τη χώρα ή το Ρουμανοπολίτη, τους Ρουμάνους πολίτες. Είναι επίκριση κατά κάποιων συγκεκριμένων πρακτικών της πολιτικής πλειοψηφίας που εκπροσωπείτε εσείς αυτή τη στιγμή και έχω κάθε δικαίωμα να το πράξω αυτό, να επικρίνω αυτές τις πρακτικές, γιατί είμαι επίτιμος πολίτης της Ρουμανικής Δημοκρατίας. Το 2001 μου ε, απονεμήθηκε, ύστερα από, την, ε, από τον αγώνα στον οποίο αποδίθηκα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί κανείς δεν μου το είχε ζητήσει να προσπιστώ τα δικαιώματα της Ρουμανίας μέσα από τη συνθήκη της Νίκαιας, γιατί κάποιοι είχαν ε, την υπέροχη ιδέα, επειδή η Ρουμανία είναι χώρα της Ανατολική Ευρώπης, να τις περιορίσουν τα δικαιώματα, τα ε, ψήφους που τις αντιστοιχούν. Και μου χορηγήθηκε η ε, ιδιότητα του πολίτη, του επιτιμού πολίτη. Γιατί μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τα ε, ίδια δικαιώματα, ισότιμα δικαιώματα λοιπόν, για το, Ρωμένο, για το Ρωμανό πολίτη. Με την προσχώρηση. Μην το δείτε λοιπόν σαν επίκριση. Ακούστε αυτό που σας λέω και ακολουθήστε αυτούς τους αγώνες. Καταστείτε γνήσια πρωθυπουργό της χώρας σας. Καθαρίστε την ε, διαφθορά και την ε, βρώμα του παρελθόντος και έρθείτε σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της διαφθοράς. Ευχαριστώ εκ μέρους των Πρασίνων, κυρία Σκά Καλώς ορίσατε κυρία Πρωθυπουργέ και η Ρουμανική Προεδρία. Καλώς να ορίσει. Πάντα είναι μια ευκαιρία να λάμψει μια χώρα η Προεδρία και να δείξει ε, τις ικανότητές τη στη διπλωματία, στους συμβιβασμού στις προόδου και να εντυπωσιάσετε και με τις δεξιότητές σα ως χώρα και ως ε, Πρωθυπουργό. Αυτό ε, είναι και βασικός μας ρόλος στις ε, θεσμικές σχέσεις και για να προχωρήσει η Ευρώπη. Αλλά η Προεδρία φέρνει και μια κυβέρνηση και μια χώρα στο προσκήνιο. Και αυτά που ανακαλύπτουμε για την ρουμανική κυβέρνηση μας ε, προκαλούν ανησυχία. Έχει μακρά παράδοση η Ρουμανία στον αγώνα για την ελευθερία και τις δημόσιες ελευθερίες. Απέταξαν μετά από 42 χρόνια μια δικτατορία οι Ρουμάνοι και η Ρουμανία έχει κάνει πολύ μεγάλες προόδους ε, κατά της διαφθοράς. Και μάλιστα οι Ρουμάνοι μπορεί να είναι περήφανοι γι' αυτό και εμείς για όλα αυτά τα επιτεύγματα του ρουμανικού λαού. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι και πάλι βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν πολιτικές ελευθερίες και χρηστή διακυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εισακούονται όμως. Αντίθετα, το η κυβέρνηση έχει οργανώσει πάταξη αυτών των ελευθεριών και των πολιτών και κατά της χρηστής διακυβέρνηση. Και τελικά ε, τίνει νομοθετικά να νομοποιήσει τη διαφθορά. Και μάλιστα ε, θα περιστελούν και οι διαμαρτυρίες. Θα πρέπει όμως μια προεδρία να δίνει το καλό παράδειγμα και να έχει και αξιοπιστία για να έχει ηγετική στάση. Έχετε ακόμα χρόνο να γίνετε το καλό παράδειγμα που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά ο χρόνος λιγοστεύει. Υπάρχουν πολλά ε, γεγονότα αυτό το εξάμεινο, το Brexit είτε έρθει είτε όχι, οι ευρωεκλογέ και ταυτόχρονα χρειάζεται και ένα όραμα μακροπρόθεσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά έχετε προγραμματίσει μια σύνοδο κορυφή το Μάιο, αλλά για να βοηθήσει αυτή η σύνοδο θα πρέπει να ασχολείται με τα φλέγοντα ζητήματα που θα πρέπει να λύσουμε. Τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή, πώ θα τη σταματήσουμε, πώ θα περάσουμε σε μια οικονομία χωρί διοξίδιο του άνθρακα, πώ θα έχουμε κοινωνικά δικαιώματα ε, που να είναι πραγματικό πραγματικότητα και όχι ωραία λόγια και πώς ε, θα ε, ε, σταματήσουμε την υποχώρηση του κράτους δικαίου σε κάποια κράτη-μέλη. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ελπίζουμε να μας εκπλήξετε θετικά. Ευχαριστώ. Μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Προεδρία της Ρουμανίας θα κληθεί να διαχειριστεί τη βαθιά οικονομική κρίση και τις τραγικές συνέπειες της τη διεύρυνση των ανισοτήτων τη συνεχή αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους και τη φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας του κόσμου χωρίς να υπάρχει ελπίδα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η στατιστική για το 2017 ένας στους 7 συνταξιούχους είναι στο όριο της φτώχειας με αυξητική τάση. όλα αυτά όλα αυτά είναι που οδηγούν και τους λαούς στη μεγάλη αφισβήτηση της ένωσης. δεν μπορεί λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση και η προεδρία σας να ζητούν την εμπιστοσύνη των λαών εν ώψη των ευρωεκλογών εάν δεν σταματήσει πρώτα η αιμονή στην πρόθεση των καταστροφικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών η στήριξη του συμφωνίου σταθερότητας η ευάθυνση της οικονομικής και δημοσιονομικής ένωσης καθώς και η λογική των προπολογισμών λιτότητας κυρία πρωθυπουργέ η gue σα σας καλεί να αφουγκραστείτε τι ανησυχίε των λαών να προωθήσετε τι θέσει των προοδευτικών δυνάμεων του κοινοβουλίου για την ανάγκη ενίσχυση τη κοινωνική πολιτική. η κοινωνική ένδυα και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων που έγινε κανόνα, επιβάλλουν να επενδύσουμε άμεσα σε ένα κοινωνικό πυλώνα ο οποίο να έχει πραγματικό περιεχόμενο στη βάση των αναγκών τη κοινωνία. γιατί δυστυχώ σήμερα αποτελεί απλά συστηματικά ευχολόγια χωρίς καμιά δεσμευτική ισχύ. πρέπει επιτέλους να προηγηθούν μέτρα και να γίνουν επενδύσεις που να δώσουν όθηση στην πραγματική οικονομία να φέρουν ανάπτυξη προς όφελος των λαών και να ενισχύσουν την κοινωνική ε, συνοχή. αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει να τεθούν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. ακόμα και η ψηφιοποίηση που τίθεται ως προτεραιότητα της προεδρίας σας πρέπει να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. εξίσου σημαντικό είναι να επιδειχθεί έμπρακτη αλληλεγγύη προ τα κράτη μέλη για μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση και όχι ενίσχυση τη λογική μια ευρώπη φρούριο. και τέλο αντί να δίνονται πακτολοί χρημάτων στην τουρκία και να τίθεται στην ημερήσια διάταξη αναβάθμιση των τολωνιακή ένωση πρέπει να ασκηθούν πιέσει στην τουρκία να σταματήσει τι πειρατικέ ενέργειε σε βάρο τη κυριαρχία των κρατών μελών όπω είναι η ελλάδα και η κύπρο στο αιγαίο και στην ανατολική μεσόγειο. ευχαριστώ πρόεδρε. E Ευρώπη των Ελευθεριών και της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Πάξας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και περισσότερα θέματα ε, με τα οποία ασχολείται. Έχουμε πολλές κοινέ αρχές και αξίες και τα συζητούμε ε, εδώ και καιρό. Τώρα έχουμε φτάσει στη φάση της εφαρμογής πολλών πολιτικών. Κυρία Πρωθυπουργέ, θα συμφωνούσατε ότι σήμερα, σήμερα το σημαντικότερο είναι να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, ε, για ποιο λόγο ε, το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ονοποίηση έχει γίνει τώρα ενδιαφέρον για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τόσοι πολλοί Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και λοιποί να μην πάρουν τον ίδιο δρόμο. Κυρία Πρωθυπουργέ, για να απαντηθούν όλα αυτά τα ε, ερωτήματα. Δεν χρειάζονται και άλλα προγράμματα για οικονομική ανάπτυξη κλπ. Χρειάζεται να αλλάξει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ομάδα των ελευθεριών της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κ. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα ε, μέχρι τώρα μου τράβηξαν την προσοχή. Πρώτον, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που έχει βάλει ε, θέμα τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων και συγχαρητήρια. Και μετά ο κύριος Μπούλμαν που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα ε, πέφτει στα παλιά πολιτικά πρότυπα και περνάει στην αντεπίθεση. Ε, αυτά είναι πράγματα παροχημένα, ανήκουν πια στην ιστορία. Τώρα αναλαμβάνεται την Προεδρία, παραδίδει η Αυστρία είναι πολύ ε, μεγάλο και φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία διότι είναι δύσκολα τα θέματα και πραγματικά διαλέξατε θέματα καθόλου εύκολα, τα ακούσαμε προηγουμένως. Εγώ εκτιμώ πολύ τη Ρουμανία και τους Ρουμάνους. Έχω όμως κάποιες αμφιβολίες αν είναι σε θέση η κυβέρνησή σας να ε, δημιουργήσει και να διαμορφώσει μια ε, λογική προεδρία και δεν ξέρω αν είστε αρκετά σταθερή κυβέρνηση, γιατί στην τρέχουσα θητεία είστε η τρίτη πρωθυπουργό. Ε, και δεν θα πρέπει να αναλωθούμε τώρα σε μάχες εξουσίας. Υπάρχει νομοθεσία ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς που προετοιμάζεται. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε όταν έρθει η ώρα. Και λήξη Προεδρία. Ο λόγος στον κύριο Ιβαν, μη εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, σε αντίθεση με όσα σχολιάστηκαν και ακούστηκαν σήμερα, πιστεύω ότι αυτή η Προεδρία θα είναι μια Προεδρία επιτυχίας. Έχω την πεποίθηση ότι η Προεδρία της Ρουμανίας θα είναι μια επιτυχής Προεδρία, γιατί χρειαζόμαστε να πετύχει η Προεδρία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή. Πρέπει όλα όσα είπαμε και συζητάμε εδώ να λάβουν χώρα. Και γι' αυτό έχετε την υποστήριξή μου. Δεν ε, μας επιτρέπει ο χρόνος παρά να αναφέρουμε δύο θέματα τα οποία εγώ θεωρώ σημαντικά. Καταρχήν, τα τρία τέταρτα των κρατών μελών αντιμετωπίζουν ε, όλο ένα και μεγαλύτερη σύγχρονη σκλαβιά στερούνται οι άνθρωποι την ελευθερία τους, εργάζονται χωρίς να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και πλήττεται όχι μόνο η Ρουμανία, αλλά στα τρία τέταρτα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντάμε αυτό το φαινόμενο. Μόνο στη Γερμανία είχαμε πάνω από 170.000 πολίτες που ήταν θύματα της σύγχρονης δουλείας. Το δεύτερο σημαντικό θέμα, μιλάμε για τη συνοχή. Σίγουρα χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους. Το άμεσο και το μέσο κόστος της διαφθοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει περίπου σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στη Ρουμανία ε, χάνουμε περίπου 40 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, πριν ήταν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ το κόστος στην Ιταλία 2 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται ΙΟΣ. Στην Ισπανία 120 δις κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα ανακτήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνοχή για την οποία μιλάτε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα στο θεματολόγιο της Προεδρίας. Καλησπέρα σε όλου. Προσκαλώ όλου του συναδέλφου να σέβονται το όριο του χρόνου, διότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Για Σούιτσα, για ένα μισή λεπτό. ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζω την εκπρόσωπο της Ορμανικής ε, Κυβέρνησης. Χαίρομαι που αναλάβατε και την Προεδρία. Έχουμε την πρώτη Προεδρία του νέου τρίου και σε αυτήν συμμετέχει και η χώρα μου, η Κροατία και είμαι πεπισμένη ότι θα συνεργαστούμε επαρκώς. Είδα προσεκτικά το πρόγραμμα εργασίας σας και είμαι σίγουρη ότι τα ζητήματα συνοχής ε, θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ. Επίσης για αυτό το οποίο είπατε για την σύνδεση και τη γεφύρωμα του καινού Βόρειας και Νότιας Ευρώπης ε, και επίσης η ασφαλή Ευρώπη την οποία αναφέρατε είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει και η Ρουμανία και η Βουλγαρία και η Κροατία να μπουν στο χώρο Σέγγεν. Ελπίζω λοιπόν να μα βοηθήσετε για να μην έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Επιπλέον στις προτεραιότητά σας ε, συμπεριλάβατε και την ισχυρή Ευρώπη που θα είναι ένας παγκόσμιος εταίρος. Βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ανησυχεί επίσης αυτό το οποίο είπατε ως τελευταίο σημείο την Ευρώπη των κοινών αξιών. Βεβαίω υπάρχουν διάφορα ζητήματα εδώ πέρα, τα ακούσατε από τους συναδέλφους, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, πολλές διαδηλώσεις, ε, δυσαρέσκεια στους δρόμους και στη Ρουμανία. Σε εσά μάλιστα ίσως ε, αμφισβητείτε και το κράτος δικαίου. Και είπατε ότι πρόκειται βεβαίως για ένα ζήτημα επικουρικότητας. Έχετε ακούσει το τι φωνάζουν οι πολίτες στους δρόμους της ε, Ρουμανίας. Τους έχετε ακούσει όντως και θα τα εφαρμόσετε αυτά τα οποία ζητάνε. Και θέλετε να υπερασπίσετε το κράτος δικαίου στην χώρα σας. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ, Ροντρίκες. Welcome, ε, ήρθατε κυρία Πρωθυπουργέ. Η Προεδρία της Ρουμανίας θα είναι η πρώτη Προεδρία της χώρας σας. Και η τελευταία πριν από Και θα ήθελα τώρα να εστιάσω στην Σύνοδο Κορυφής του Σιμπίου που είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να παρουσιάσουμε μια άλλη Ευρώπη για όλους τους πολίτες στην Ευρώπη πριν από τις ευρωεκλογέ. Να σας πω λοιπόν τι προσδοκούμε εμείς από εσάς για το τι είδους Ευρώπη θέλουμε εμείς μέσω της ε, Συνόδου Κορυφής του Συμπίου. Θεωρούμε ότι έχετε τις σωστές προτεραιότητες για να έχουμε ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων, συνοχή και οπωσδήποτε εδώ πέρα ε, η συνοχή είναι η λέξη κλειδί. Όπως είπατε, οικονομική, κοινωνική, πολιτική συνοχή. Είμαστε στο πλευρό σας. Και βεβαίω μπορεί να γίνει κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Ο κοινωνικός πυλώνας να γίνει ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεύτερον, μία πρώτη συμφωνία για τον πολιετή προϋπολογισμό όπου θα έχουμε ως κύρια ανησυχία την συνοχή. Θα περιλαμβάνει τα κρατη και την Ευρωζώνη. Και βεβαίως, ναι, να έχουμε μια Ευρώπη που θα βασίζεται στα ε, ευρωπαϊκά σύνορα και με την Ρουμανία. Το πρώτο είναι ακριβώς αυτή η συνεργασία με όλες τις σχετικές ε, χώρες. Το περιλαμβάνει και την ανατολική εταιρική σχέση που σας απασχολεί πάρα πολύ. Και βεβαίως αν τα καταφέρουμε σε αυτό θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τη μετανάστευση. Και τέλος, ε, αν έχουμε αυτήν την Ευρώπη, θα έχουμε και ενότητα εότι και αν γίνει ιστορικό λοιπόν καθήκον, αλλά και μια ευκαιρία που έχετε. Ο κύριος Ντίβα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Ρουμανική Προεδρία είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει, είμαστε σε καλά χέρια για το Brexit. Θέλω να μας βοηθήσετε σε αυτό. Πριν από δύο χρόνια θεωρούσαμε ότι θα είναι κάτι εύκολο το Brexit. Σήμερα είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουν να ξεφορτωθούν. Και είναι δύσκολα τα πράγματα για την Πρωθυπουργό, την κυρία Μέη, η οποία πραγματικά έσφιξε τα δόντια και κάνει ό,τι μπορεί. Στη Βουλή των Κοινοτήτων απόψε θα γίνει χαμός. Αλλά βεβαίως η Πρωθυπουργό μας ε, δεν θα αλλάξει πορεία στη μέση του δρόμου. Ξέρει πως τα πράγματα είναι ζόρικα, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για την Βρετανία. Βρίσκεται βεβαίω μεταξύ σφυρας και άκμονος, αλλά αναμένουμε με κομμένη την ανάσα για κάποια επιτυχία. Ο κύριος Ζαντόφσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχηθώ ιδιαίτερα αποτελεσματική προεδρία στην Ρουμανία. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, τους ε, νέους σχεδιασμούς της μεταναστευτικής πολιτικής, Υπάρχει μια σειρά δράσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Επίσης, η πολιτική συνοχή αποτελεί προτεραιότητα, πολύ σημαντική για μένα και είμαι σίγουρος ότι η Ρουμανία θα δώσει μια γεωπολιτική χρειά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και στα ανατολικά της Επίρου μας και σε σχέση με τη Ρωσία. Βέβαια, οι κύριες αξίες, ο σεβασμός ε, του κράτους δικαίου είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε στη Ρουμανία να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια. Υπάρχει μια ερώτηση για σας, δέχεστε, παρακαλώ, κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναμφισβήτητα, η εκπεριτροπής Προεδρία θα είναι μια προκλητική Προεδρία. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για το μέλος της Ευρώπης ε, όταν ε, παράλληλα τρέχει το Brexit. Όμως είναι πολύ εύκολο για κάποιους να μιλούν εκτός πραγματικότητας. Και αυτή η παραπληροφόρηση και η έλλειψη συνοχής ε, στο να κάνουν κάποιες δηλώσεις ε, είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφισβήτητα το κράτος δικαίου αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρουμανία και αυτό το φαίνεται... Πρέπει να κάνετε μια ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Μια ερώτηση πρέπει να θέσετε στον προηγούμενο μιλητή, στον κύριο Βιονταστόφσκι. Είμαστε δύο νικολάοι, κύριε Πρόεδρε. Ποιο μπορεί να μιλήσει. Ζητήσατε το λόγο. Για μπλε κάρτα. Θέλετε να θέσετε μια ερώτηση. Okay. Euh, Αν δεν έχετε ερώτηση, όχι, δεν έχω ερώτηση. Και ε, μετά θα σας δώσουμε το λόγο τότε. Ε, Ο κύριος ε, Χόκμαρκ, παρακαλώ, για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι είναι φανταστικό το ότι η Ρουμανία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σημάδι για το πώς ε, έχει αναπτυχθεί η Ευρώπη όμως σίγουρα θα είναι φανταστική η εξέλιξη και θέλω να πω ότι εσείς και η δική σας κυβέρνηση πρέπει να καταπολεμήσετε τη διαφθορά όπως απαιτούμε και από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το να συγχωρείτε διεφθερμένους πολιτικούς επειδή λέγεται ότι είναι, υπάρχει υπερπληθυσμός στις φυλακές δεν είναι αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να καταπολεμάτε όσους καταπολεμούν τη διαφθορά είναι απαράδεκτο. Η αποποινικοποίηση της διαφθορά. η, η αμνίστευση διαφθαρμένων για να προστατεύσετε τους δικούς σας δεν είναι αποδεκτό. Άκουσα ότι ο Ντο Μπούλμπαν σας υπεράσπισε, ο επικεφαλής σοσιαλιστικής ομάδας. Όμως αυτό είναι ντροπή για τη σοσιαλιστική ομάδα, πρέπει να πω. Υποτίμησε τον εαυτό του και εσείς θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη να προστατεύσετε τη Ρουμανία γιατί πιστεύουμε ότι είναι φανταστικό το ότι έχετε αναλάβει την Προεδρία αλλά μην τα θαλασσώσετε. Έχετε μια ευθύνη και πρέπει να την αναλάβετε. Κύριε Χόκμαρκ, υπάρχει μπλε κάρτα για σας, δέχεστε? Από τον κύριο Φρουντσουλίκα, παρακαλώ, η ερώτησή σας. αγαπητέ συνάδελφοι. Δεν πιστεύετε ότι είναι ντροπή σήμερα ο πρόεδρος ε, του ΕΛΚ, ο κύριος Σοζουφτόλ, συνεχάρει τον κύριο Γιωχάνης και του είπε ότι θα ε, υλοποιήσει μια εξαιρετική προεδρία όταν ξέρουμε όλοι ότι η εκπεριτροπή προεδρία του Συμβουλίου την αναλαμβάνει η κυβέρνηση της Ρουμανίας και επικεφαλής είναι η Ρουμάνα Πρωθυπουργός. Δεν είναι λοιπόν ντροπή ο κύριος Κούρς στις 21 Δεκεμβρίου του Βουκουρέστη, στο Βουκουρέστι παρέδωσε συμβολικά την Προεδρία του Συμβουλίου στον πρόεδρο Γιωχάνη, κάνοντας εκ νέου ένα μεγάλο πολιτικό λάθος. Και ταυτόχρονα ε, ουσιαστικά παραπλάνησε τους πολίτες που πρέπει να ξέρουν την αλήθεια. Παρακαλώ να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κάπου έφυγε εκτός θέματος ο συνάδελφος, γιατί εγώ μιλούσα για τα προβλήματα της διαφθοράς στη Ρουμανία. Όπως ε, μας έχει καταδείξει η Transparency International, η Επιτροπή της Βενετίας και πολλοί άλλοι. Και το γεγονός της αμνίστευσης ε, διεφθαρμένων πολιτικών και μόλις μίλησε ο υπουργό ε, στο BBC. Είπατε ότι κάποιοι δίνουν τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο της χώρας σας. Ε, τι να σας πω, εμένα δεν με ανησυχεί και πολύ αυτό. Νομίζω ότι εσείς και οι σοσιαλιστές εδώ θα πρέπει να, είναι, να είστε τόσο αυστηροί με τη Ρουμανία όπως είμαστε και με την Ουγγαρία ή την Πολωνία. Γιατί η κατάχρηση εξουσίας πάντοτε είναι κατάχρηση εξουσίας. Θα πρέπει και εσείς και εμείς να την καταπολεμήσουμε. Κυρία Φαγιόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, στην αρχή της Προεδρίας σας έχετε προσελκύσει ήδη μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ωστόσο ότι θα πετύχετε τους στόχους σας στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Εγώ σας υποστηρίζω, ιδίως ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να δείξουμε θετική θετικά παραδείγματα ε, σε αυτήν την περιοχή της Ευρώπης και γι' αυτό ε, συγχαίρω τους φίλους μας ε, στην Μακεδονία που ψήφισαν υπέρ των συνταγματικών αλλαγών. Και η Ελλάδα πιστεύω ότι θα ψηφίσει θετικά. Ήταν πραγματικά τολμηρό και σοφό εκ μέρους των ηγετών να επιδιώξουν την επίλυση αυτής της διαφιλονικίας. Καλό λοιπόν τους ηγέτες της περιοχής και την Προεδρία να εξομαλύνουν με μεγάλη αυστηρότητα ε, την κατάσταση. Να μην υπάρχει μίσο και καχυποψία κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χρειαζόμαστε ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα έχει και κοινωνική διάσταση. Θέλουμε να είναι σταθερή και ειρηνική. Εύχομαι να οδηγήσετε εσεί την Ευρώπη σε αυτή την πορεία. Ευχαριστούμε. Τόμας, έτσι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ρουμανία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα διάστημα χρονικό ιδιαίτερα δύσκολο. Θα πρέπει να επικεντρωθείτε στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και να λάβετε υπόψη και την απώλεια ενό του κράτου μέλου, μαζί με τι ευρωεκλογέ που θα καθορίσουν το μέλλον τη Ένωσή μα. Ελπίζω λοιπόν ότι τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρουμανία δεν θα πλήξουν και τι φιλοδοξίε τη, όπω τι έχει εκφράσει στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χάσει χρόνο, διότι για να επικεντρωθούμε στι οικονομικέ μα προτεραιότητε θα πρέπει να βιαστούμε. Ούτε τι μεταναστευτικέ προκλήσει μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αργότερα, γιατί από εμά περιμένει μια ε, θαραλέα κίνηση ο υπόλοιπο κόσμο. Ελπίζω λοιπόν η Ρουμανική Προεδρία να ε, ασχοληθεί με την επίλυση αυτών των προβλημάτων όπω έχει ανακοινώσει. Και η ασφάλεια δεν θα πρέπει να ε, γίνει μια ε, πουσιώδη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ασφαλή όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό το αποδεικνύουν οι πολλαπλέ απόπειρε. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των προτεραιότητων μα. Ο κ. Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα να μπορώ να διαπραγματεύομαι τα νομοθετήματα με την Ρουμανική Προεδρία. έχω την εξή θέση ως μέλος του ΕΛΚ. Εργάζομαι ήδη και θα εργαστώ με τη μόνιμη προσωπία της Ρουμανίας και θα συνεισφέρω στο να κλείσουν νομοθετικοί φάκελοι. Θα συνεχίσω να υπερασπίζω τα συμφέροντα των Ρουμάνων σε όλου τους φακέλους που είναι σε εξέλιξη. Δεν δέχομαι θέσεις ε, ε, κατά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και εγώ θα θα καταφερθώ κατά θέσεων που αφορούν τον περιορισμό της κυκλοφορίας των εργατών. Κυρία Ντανσίλα, Μιλήσατε πολύ για την πολιτική συνένεση σε εσωτερικό επίπεδο. Εγώ δεν ε, συμφωνώ με τέτοια συνένεση κατά των ευρωπαϊκών αξιών του κρατούς δικαίου και της δικαιοσύνης. Ε, ζητήσατε ένταξη στο χώρο Σενγκεν. Δεν είναι πολύπλοκο. Διορθώστε τους νόμους περί δικαιοσύνης. Ε, στείλετε τους υπουργού να συζητήσουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε και να πείσουν τις κυβερνήσεις να ψηφίσουν υπέρ της Ρουμανίας. Και ε, όποιον στείλετε θα προεδρεύσει και του Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Χρησιμοποιήστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ρουμανία χρειάζεται νοσοκομεία, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές. Αν κάνετε όλα αυτά θα δείξετε ότι είστε στην πλευρά των Ρουμάνων και θα κερδίσετε το σεβασμό των Ευρωπαίων εταίρων. Η υποχρέωσή σας είναι να εκπροσωπήσετε τη Ρουμανία σύμφωνα την επιθυμία της ε, πλειοψηφίας ε, των πολιτών και όχι σύμφωνα με την πλειοψηφία των βουλευτών ε, του. Έχετε μία μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Ο κύριος Γιάκον Σάρη, παρακαλώ, κάντε την ερώτηση. Η κυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναρωτιόμουν για το ότι κανείς δεν μίλησε για μία από τις ε, μεγαλύτερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη που λαμβάνει η χώρα στη Ρωμανία, δηλαδή τους Ρωμά και τη μεταχείρισή τους. Και εσείς ε, είστε Πρωθυπουργό, Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω μήπως αυτό οφείλεται ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή συχνά σε τέτοιες συζητήσεις είμαστε τόσο ευγενικοί και δεν θίγουμε τα δύσκολα. Σας ευχαριστώ ο κύριος Μαρινέσκου για να απαντήσει. Είναι μία ερώτηση που προέρχεται από έλλειψη σωστή ε, ενημέρωση. Ε, Σα καλώ να έρθετε στη Ρουμανία και στη δική μου περιφέρεια, όπου ήρθαν ε, και άλλοι συνάδελφοι, να επισκεφτείτε την πόλη και την περιοχή σας. Καλό να έρθετε και να δείτε τι συμβαίνει σε σχέση με το θέμα που θίξατε εδώ στη Ρουμανία. Ευχαριστούμε ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Γιώζεφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρωθυπουργέ, κάθε χρόνο αλλάζει η Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι δηλαδή κάτι το σύνηθες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάληψη της ε, Προεδρίας από τη Ρουμανία αποκλίνει αυτό το, αυτό το σχήμα γιατί αφενός ε, υπάρχει ιδιαίτερη χρονική πίεση και από την άλλη ε, όλη η χώρα πλέον ε, είναι υπό το μικροσκόπιο ολόκληρης της Ευρώπης. Ε, η Κομισιόν πριν από λίγες εβδομάδες διαπίστωσε μια στασιμότητα όσον αφορά την κατάσταση του κράτους ε, δικαίου στην χώρα. Η Ρουμανία λοιπόν θα βρεθεί υπό το μικροσκόπιο του επόμενου μήνε. Και εδώ πέρα υπάρχει μια ευκαιρία. Η χώρα μπορεί να δείξει ότι είναι ικανή να επιλύσει τα εσωτερικά τη προβλήματα και τι υποχρεώσει ε, που έχει. Είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να επιτύχει πολλά η Ρουμανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα σα στηρίξουμε σε αυτό. Σα ευχαριστώ, Γιώζεφ. Κύριο Γιούρεκ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν να χρησιμοποιήσω το λεπτό μου θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μπούλμαν πριν 20 λεπτά παρενέβη. Εγώ τότε είχα ζητήσει να πάρω το λόγο γιατί ήθελα να αφιστήσω την προσοχή του Προέδρου Ταγιάννη. Το άρθρο 11 του κανονισμού μας υποχρεώνει στο να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και να μην προβαίνουμε σε δηλώσεις δυσφημιστικές. Τώρα, πρόκειται για μια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε ως φασιστική. Ε, εδώ μιλάμε για ε, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες αυτού του κοινοβουλίου να επιτίθεται σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι παραδεκτό αυτό. Ο πρόεδρος έπρεπε να έχει αντιδράσει αμέσω. Και όταν ένας βουλευτής ζητά το λόγο, δεν ε, είναι δυνατό να μην δίνεται το λόγο για ένα διαδικαστικό ζήτημα. Ο κύριος Μπούλμαν δεν είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να αντιδρά στις παρεμβάσεις άλλων συναδέλφων. Γι' αυτό εγώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή, προσοχή του Πρόεδρου Ταγιάννη στο γεγονός αυτό. Τώρα, σε σχέση με την απάντηση του κυρίου Μπούλμαν, δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά του Προέδρου και Τώρα να περάσω και στη δική μου παρέμβαση. Τώρα αρχίζει να μετράει το δικό μου λεπτό. Συγγνώμη. Εσείς πήρατε το λόγο για ένα θέμα που έχει να κάνει με τον πρόεδρο Ταγιάννη που ήταν εδώ στην αίθουσα και ξέρει πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Εγώ θα του το παραπέμψω. Όμως αυτό έχει να κάνει με τη δική του παρέμβαση. Παρακαλώ. Κύριε Σαντρία, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Ήθελα να μιλήσω σήμερα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με την ευκαιρία τη επισκεψή σα. Όπω ξέρετε, η θέση του Κοινοβουλίου εδώ είναι ξεκάθαρη. Χρειάζεται ένα επίπεδο δαπανών φιλόδοξο, το οποίο να ασχολείται με την υλοποίηση των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη, ξεκινώντα από την καταπολέμηση τη ε, υπερθέρμανση του πλανήτη και των κοινωνικών ανισοτήτων καθώ και των εδαφικών. Ε, εδώ βλέπουμε να αναδαβλίζονται, οι, οι εξτρεμισμοί, να κινδυνεύει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και η οικονομική μα σταθερότητα. Θα πρέπει το Συμβούλιο να καταλάβει ότι χωρί αυξήσει στου ίδιου πόρου, το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να δώσει τη συνένεσή του για την διάσταση των δαπανών. Θα πρέπει λοιπόν και για του πόρου να δείτε ότι είναι μηδενική η πρόοδό μα. Θα πρέπει να δούμε τι αδρέ γραμμέ ε, πιθανή συνεννόησή μα για τι ε, δημοσιονομικέ γραμμέ. Τι εννοείται από τη μια μεγάλε γραμμέ και από την άλλη πώ θα λάβετε υπόψη τι διαφορετικέ θέσει του Κοινοβουλίου στα διάφορα αυτά θέματα. Ευχαριστούμε, κυρία Μπρέσο. Παρακαλώ, Μερτσέντε, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, και από μένα πολλέ ευχέ για καλή έκβαση στην Προεδρία σα. Ευχαριστούμε για τις τέσσερις θεματικές προτεραιότητες που μας ε, αναφέρατε. Θέλω να σχολιάσω το θέμα της εδαφικής σύγκλησης. Πιστεύω ότι καμία περιοχή της Ευρώπης, όπως θυμήσατε κι εσείς, δεν πρέπει να μείνει ε, καθυστερημένο στην ε, πρόοδο που θα κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί, ε, όπως είπαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από κάποιο καιρό, Χρειάζεται ένα κατάλογο προτεραιοτήτων και για τι περιοχέ που έχουν καθυστερήσει αυτέ τι υπαίθρου, τι ορεινέ και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Όχι μόνο λοιπόν για τι αστικέ περιοχέ, αλλά και για αυτέ τι ε, απομακρυσμένε περιοχέ, τι μειονεκτούσε περιοχέ. Κατάλογο προτεραιοτήτων. Το έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο με μια πρωτοβουλία του. Πρωτοβουλία που ξεκίνησε μια πρώτη μελέτη του θέματο και θα μπορούσε μετά να οδηγήσει και σε εκπόνηση μια ε, τέτοια ε, ιεραράχηση των στόχων. Είναι σημαντικό λοιπόν η Προεδρία, γιατί η Ρουμανία είναι μια χώρα με πολλέ ε, περιοχέ υπαίθρου, αγροτικέ περιοχέ, ορεινέ περιοχέ στην Ευρώπη. Τα γνωρίζετε καλά. Ε, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στι ευρωεκλογέ φέτο. Τι σκέφτεστε να κάνετε για να συμμετάσχουν ενεργότερα και για να του εξυπηρετήσετε και να του βοηθήσετε μάλλον και να διευκολύνετε την έλευσή του στι κάλπε. Ευχαριστούμε κύριε Μπρέσο, κύριε Μπρέσο, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητά μέλη της κυβέρνησης, καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ που παρουσιάσατε τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Και επίσης ε, θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να μην μπερδευτείτε εδώ, επειδή το τι είπε κάποιος συνάδελφος εδώ δεν είχε καμία σχέση με την Προεδρία της Ρουμανίας, ούτε με το πρόγραμμα με των δραστηριοτήτων απλώ εντάσσεται στην προεκλογική εκστρατεία. Θα πρέπει να κατανοήσετε τον κύριο Βερχόφστατ. Ε, ε, δεν ε, φτάνει το αντίστοιχο κόμμα στην Ρουμανία στο εκλογικό κατόφλι και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ταυτόχρονα θέλω να σα ενθαρρύνω μαζί με του 200 υπαλλήλου τη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ρουμανία μαζί και με άλλου εκατοντάδε υπαλλήλου που στη Ρουμανία προετοιμάζουν την Προεδρία. Να ακολουθήσετε το χρονοδιάγραμμα παρουσίας σας κυρία Πρωθυπουργό, γιατί οι τέσσερις πυλώνες, η σύγκληση, η ασφάλεια, η παγκόσμια Ευρώπη και η Ευρώπη των αξιών είναι ένα θέμα που θα μείνει στη Ρουμανία, στην ιστορία για τη Ρουμανία και θα θεωρηθεί ότι είναι το πιο πολιτικό σημαντικό βήμα που έκανε η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και καλή επιτυχία κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ κυρία Νίκα. Η κυρία Τόια, παρακαλώ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, θέλω να χαιρετήσω την Πρόεδρο του Συμβουλίου σε αυτό το στάδιο. Είναι μια συνάδελφος που την εκτιμούσαμε στην ομάδα μας και στο Κοινοβούλιο. Θέλω να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές γιατί αναφέρθηκαν πολλά από τους συναδέλφους της ομάδας μου και θέλω να αναφερθώ σε δύο σημαντικές στο θέμα του κοινωνικού πυλώνα είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες ε, που παρουσίασε στο πρόγραμμά της η Ρουμανική Προεδρία και νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα θέμα αξιολόγηση της δράσης και της ικανότητας της Ευρώπης σε αυτή την κρίσιμη εποχή για τους Ευρωπαίους πολίτες σε κάποιες ε, χώρες είναι πιο προφανής η κοινωνική προσοχή ε, που, της οποίας χρήζουν οι πολίτες μας, σε άλλες δεν είναι τόσο προφανής, όμως χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να ε, φροντίζει τα παιδιά και να προωθεί την ευημερία. Μία άλλη πτυχή είναι αυτή της βιομηχανίας. Εγώ τα βλέπω μαζί, γιατί μια Ευρώπη που μεγενθύνεται είναι και μια Ευρώπη που μπορεί να είναι πιο κοντά στις ε, ανάγκες και σκέφτομαι και το πρόγραμμα Ορίζοντα, Horizon και εγώ νομίζω ότι η Προεδρία θα πρέπει να ολοκληρώσει με τη συνεισφορά όλων. Σας ευχαριστώ και καλή δουλειά ο κύριος Ντάντη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, Καλώ επιστρέψατε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, την αίθουσα τη Ολομέλεια. Δεν έχετε πολύ χρόνο λόγω των ευρωεκλογών. Θα πρέπει να ασχοληθείτε με σημαντικά θέματα. Νομοθετική δουλειά σημαντική μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο. Επειδή δεν υπάρχει πολλή χρόνο, θα σταθώ σε ένα σημείο που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Το θέμα τη ενιαία αγορά. Όπω όλοι ξέρουμε, είναι μια μεγάλη, από τι μεγάλε επιτυχίε τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δυστυχώ όμω έχει ακόμα πολλέ αδυναμίε. Και τα τελευταία χρόνια έχουν ε, υπάρξει φόβοι λόγω της ενίας αγοράς και αντιευρωπαϊκές τάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη οδό δράση, πορεία δράση μάλλον, με κανόνε αυστηρού για την ψηφιακή μετάβαση τη ε, κοινωνία και τη οικονομία μα. Και επ' αυτού να υπογραμμίσω το εξή. Ένα ακόμη θέμα τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς. Ελπίζω μαζί με την Ρουμανική Προεδρία να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τις διαγματεύσεις της προσεχής εβδομάδες. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες προϊόντα ασφαλή ιδίω αυτά που πολλούνται στο διαδίκτυο και σύμφωνα όλα με τα πρότυπα και του κανόνε μα. Είναι σημαντικό για την εσωτερική αγορά και για να υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων τη Επίρου μα. Ευχαριστούμε κύριε Ντάντη. Και τώρα για την διαδικασία Catch έχουμε 25 εγγεγραμμένου. Είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλου. Θα δώσω το λόγο σε 10 ομιλητέ. Ανά ομάδα για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Κύριο Πασκού. Ένα λεπτό. Κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Κάθε Προεδρία θα πρέπει να δράσει πάνω σε τρεις γραμμές. Καταρχήν να συνεχίσει τις εργασίες της προηγούμενης Προεδρίας, δεύτερον να πετύχει τους δικούς της στόχους και τρίτον να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντίστοιχη στιγμή. Μας παρουσίασε το πρόγραμμα Ρουμανία, σε σεβόμενοι αυτά τα αιτήματα. Σήμερα, όταν ε, η φιλεύθερη τάξη ε, βρίσκεται σε κρίσιμη στιγμή, η Ρουμανία προτείνει μέσω της Προεδρίας της να ενδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κύριο πυλώνα του συστήματος αυτού. Ταυτόχρονα, να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ισχυρή όχι μόνο ω ε, θεσμός αυτό καθ' αυτός, αλλά και χάρη στις προσπάθειες του κάθε κράτους μέλου Στο σημερινό κόσμο και στον ευριανό κόσμο η προστασία που προβλέπεται από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να διπλασιαστεί και να υπάρχουν και οικονομικές και στρατιωτικέ προσπάθειε από τα κράτη-μέλη παράλληλα με τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτούς τους ε, στόχου. Ε, ε, δεν μπορούμε να τους πετύχουμε μέσω της διάκρισης και την απομόνωση παρά μόνο αν υπάρχει ειλικρινή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριο Μουρεσάν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάληψη τη Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά είναι ιστορική στιγμή για τη χώρα μα και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η Προεδρία αυτή ανήκει καταρχήν στο ρουμανικό λαό. Και θέλω να πω επίση ξεκάθαρα, ο ρουμανικό λαό είναι έτοιμο για αυτή την πρώτη Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι εδώ και δύο χρόνια διαδηλώνουν οι Ρουμάνοι είτε στο δρόμο για να υπερασπίσουν το κράτο δικαίου και μια ανεξάρτητη τη δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές αξίες και το κάνουν κρατώντας ε, την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως ε, ε, πέρα από το ότι αποτελεί τιμή αποτελεί και ευθύνη η Προεδρία και εσείς κυρία Πρωθυπουργή θα έχετε την δυνατότητα να διαχειριστείτε κάποια σημαντικά θέματα. Καταρχήν, τον προπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια. Στου ε, δικαιούχου ε, θα πρέπει να δώσουμε βεβαιότητα ω προ τα ποσά ε, και ω προ τι προποθέσει βάσει των οποίων θα λάβουν χρήματα. Για τον Brexit θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει απόψε και θα πρέπει να προσφέρουμε στα εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε που βρίσκονται στη Βρετανία βεβαιότητα για το μέλλον του. Τρίτον, η Ρουμανία έχει την ε, δυνατότητα ε, να θέσει την ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως πρέπει να σέβεστε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο περιμένει και ο ρουμανικός λαός. Σας ευχαριστώ. Προσπαθήστε να σεβέστε το χρόνο, συνάδελφοι. Ο κύριος Μαριάς, για ένα λεπτό. Κυρία Πρωθυπουργέ της Ρουμανίας, εγώ θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό γιατί είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές με το συμβούλιο να είναι ανίκανο να αναλάβει τις ευθύνες του καθώς συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεχίζουν το business as usual και αρνούνται να αλλάξουν το δουβλίνο τρία που έχει μετατρέψει την ελλάδα και την ιταλία σε αποθήκες ψυχών. η ελλάδα δεν αντέχει πλέον άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. τα νησιά του αιγαίου έχουν βουλιάξει από τους μετανάστες και από τις αυξημένες ροές οι οποίες πλέον υπάρχουν και χερσαία στον εύρο. η περίφημη αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής ένωσης παραμένει γράμμα κενό. πρέπει λοιπόν να εκτελεστεί η μετεγκατάσταση. είχε εκτελεστεί μόνο κατά το. 30%. προτείνω να αλλάξει το σύστημα χορήγησης ασύλου να καταργηθεί το δουβλίνο τρία και η ρύθμιση του κράτους πρώτης εισόδου να γίνει κατανομή των αιτήσεων ασύλου καθώς και των προσφύγων και μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών με βάση την έκταση τον πληθυσμό και το αεπ. έτσι θα εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. περιμένουμε μέτρα από την προεδρία σας. ευχαριστώ. κυρία Κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω όσους εκφράσατε την εμπιστοσύνη σας στην Ρουμανική Προεδρία και εγώ ήμουν μέρος της κυβέρνησης. Ξέρω πολύ καλά τα μέλη της κυβέρνησης και είμαι σίγουρη γιατί θα ασκήσουν μια καλή Προεδρία. Για πρώτη φορά είχαμε ένα διευρυμένο συμβούλιο και εμείς ε, εργαστήκαμε ως Ευρωβουλευτές για το πρόγραμμα. Έχουμε Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά, όμως είναι λυπηρό που οι συνάδελφοί μας ε, που ήρθαν στο Κοινοβούλιο με ψευδείς πληροφορίες ε, όταν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να εξελίψουμε τις ευθύς ειδήσει. Ε, εντάξει, είμαστε τη προεκλογικής εκστρατείας, αλλά δεν πρέπει να επιτεθόμαστε σε ένα κρατός μέλος που αναλαμβάνει την Προεδρία. Πρέπει να μιλήσουμε για την προτεραιότητα, για το πρόγραμμα. Θα ήθελα να ρωτήσετε περισσότερο τι μπορούμε να κάνουμε κάνουμε, να προτείνετε προτεραιότητε. όχι να αρχίσουμε να μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε και σα διαβεβαιώ ότι δεν τα ξέρετε. Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία και μάλιστα σήμερα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια ένα θέμα για το οποίο είμαι η και θα ξεκινήσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσει. Θα δείτε τι καλή Προεδρία λοιπόν θα ασκήσει η Ρουμανία. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. κυρία Κούνεβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Το 2018 συμμετείχατε ως Ευρωβουλευτής στην εκδήλωση που διοργανώσα με δύο συνάδελφους από την πολιτική σας ομάδα, τον κύριο Πυρίνσκι από τη Βουλγαρία και την κυρία Γραπίνη από τη Ρουμανία, για να αναζητήσουμε νέους δρόμους συνεργασίας στα Βαλκάνια. Ελπίζω ότι τώρα θα πράξετε τα μέγιστα για να προχωρήσει η βαλκανική συνεργασία. ανησυχούμε όμως όταν ακούμε ότι η ρουμανία είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τις εργασιακέ σχέσει, τους μισθούς την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα. είναι έτσι; τέσσερα χρόνια δουλέψατε μαζί μα και ξέρετε τι προτεραιότητε που έχει το ευρωκοινοβούλιο κοινωνικό πυλώνα ανθρώπινα δικαιώματα αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου. αυτέ πρέπει να είναι και οι δικέ σα προτεραιότητε. σα εύχομαι καλή προεδρία και να πάνε όλα με τον καλύτερο τρόπο. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Γιάροκ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Γιάροκα. Ε, κυρία Πρωθυπουργέ, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Προεδρία σα και σα ευχαριστούμε που τονίσατε τα κυριότερα σημεία. Ένα από τα σημαντικότερα για εμά είναι η συνοχή την οποία αναφέρατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο όταν μιλάμε για τι οικονομικέ διαφορέ, όπω είπατε α, μεταξύ των ανθρώπων αλλά και την πρόσβασή του στα δικαιώματα ω Ευρωπαίοι πολίτε. Η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και αναμένουμε από εσάς να κάνετε κάτι τους επόμενους έξι μήνες γιατί θεωρούμε ότι έχετε μεγάλη πείρα σε αυτά τα θέματα. Ε, ε, έχετε, είστε σε ένα από τα πιο φτωχά κράτη-μέλη. Προσπαθείτε να αλλάξετε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση για τους Ρωμά και την απάντηση κύριε Μαρινέσκου γιατί ξέρω γιατί υπόθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναδούμε το θέμα των φτωχών. Νομίζω πως η Προεδρία σας πραγματικά πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στην Ευρώπη πως ε, υπάρχουν 220 εκατομμύρια φτωχοί στην Ευρώπη που πρέπει να βοηθηθούν. Ελπίζω λοιπόν η Προεδρία σας να προωθήσει το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ζωάνα παρακαλώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρο, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητά μέλη, της κυβέρνηση Ρουμανίας, αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως να μην είναι τυχαίο σήμερα ότι 12 χρόνια μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευκαιρία της παρουσίασης των προτεραιοτήτων ε, της ε, Προεδρίας γιορτάζει δύο σημαντικέ επαιτίου σε Ρουμανία 116 χρόνια από το γέννηση του Μιχαέ Μινέσκου, του εθνικού μας σπίτι που έχει μεταφραστεί σε πάνω από 60 γλώσσες και την ημέρα ε, του εθνικού μας πολιτισμού. Για μας αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, η Ρουμανία μέσω της φωνής της κυρίας Δαντσίλα της, της Πρωθυπουργού παρουσιάζει το όραμά της ε, για την εντολή της Προεδρίας ε, αποτελεί μια τρίτη αιτία γιορτής. Μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι γη και κόρες αυτής της μεγάλης οικογένειας. Και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην κυρία Νταντσίλα και στα μέλη της ρουμανικής κυβέρνησης και να παρακαλέσω τους συναδέλφους να έχετε εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στο όραμα της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Και για μένα είναι τιμή να εργαστώ σε θέματα που, ε, στα οποία θα εργαστεί η δική μου χώρα, έχοντας την Προεδρία. Ξέρω ότι η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη και γι' αυτό σας ρωτώ, κυρία Πρωθυπουργέ, ποιο είναι το όραμα της Προεδρίας της Ρουμανίας και τι προτείνει η Προεδρία σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, κυρία Πρωθυπουργέ, του τελευταίου μήνε και εσείς και μέλη τη κυβέρνησή σα, άσκησαν κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίξατε επανειλημμένα ότι η δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής βασίζεται σε παραπληροφόρηση και σε επιπολαιότητα. Επίση, και ε, απευθύνεται κριτική στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπατε ότι ξένες δυνάμεις ε, ε, το χειραγώγησαν και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο θεσμικούς εταίρους αφού είπατε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο και το είπατε και στους Ρουμάνους. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Τη στιγμή που εσείς συζητάτε για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στη Ρουμανία ένα τηλεοπτικό κανάλι διέκοψε την εκπομπή του γιατί. Ε, τόλμησε να δείξει εικόνες από τη διαδήλωση της 10ης Αυγούστου και είπατε, ε, όπως είπε και ο κύριος Μπουλμέν, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία στη Ρουμανία. Θα πρέπει να σε ανησυχεί αυτό, κυρία Πρωθυπουργέ αν δεν ήσασταν σε μία λογική του Τσαουσέσκου και αν δεν θέλετε να επιστρέψετε στο χρόνο, οπότε η προπαγάνδα ήταν προτιμότερη της αλήθειας ε, και κόβετε το μικρόφωνο του μιλητή. Παρακαλώ, κύριος Ρόνεν, για ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που η Ρουμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου και υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στα οποία θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο του επόμενου μήνε. Θέλω να τονίσω το θέμα τη οδηγία για την προστασία των καταγγελόντων και είτε αυτοί προέρχονται από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν κανόνε προστασία του. Θα πρέπει να μπορούν να καταγγείλουν τα δικαιώματα ή εγκλήματα που γνωρίζουν. Εάν δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ε, προστασία που θα του προσφερθεί, δεν θα περάσουν σε καταγγελίε. Το Συμβούλιο έχει αμφισβητήσει τη νομική βάση της οδηγίας. Όμως, ε, οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμφωνούν. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμένουμε σε ένα τέλμα στο Συμβούλιο. Ελπίζω ότι η Ρουμανία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της θα κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει με θετικό τρόπο τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ώστε οι καταγγέλλοντες να έχουν ευρωπαϊκή προστασία με ελάχιστα πρότυπα. Ευχαριστούμε και τώρα... Πού πήγαμε. Κυρία Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ανάληψη τη Προεδρία από τη χώρα μου αποτελεί πολύ σημαντική στιγμή για τη Ρουμανία και θα αποδείξει η Ρουμανία την διοικητική της ικανότητα και την αξία της, καθώς και το σημαντικό ρόλο που θα παίξει στην διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων και στην ε, οικοδόμηση του μέλλοντος. Θα έχει στρατηγική θέση και θα αποτελέσει ένα δεσμό που ε, θα εναρμονίσει τα διάφορα συμφέροντα που έχουν διαιρέσει την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι σημαντικότερο παρά ποτέ σε αυτή την περίοδο της γεμάτη προκλήσεις να δείξουμε ενότητα και αλληλεγγύη για το καλό των Ρουμάνων. Λυπάμαι που σα λέω κύριε Φερχόφστατ, κυρία Κέλλερ και σε άλλου που πήραν το λόγο σήμερα ότι πλανά στα ικτρά. Είναι λανθασμένες οι πληροφορίες σας ε, και σας έχουν παραπλανήσει ε, και είναι λυπηρές οι επιθέσεις που κάνετε σήμερα στη Ρουμανία και στην κυβέρνησή της ε, γράφοντας τη λογική προεκλογικής εκστρατεία. Η Ρουμανία είναι κράτος δικαίου και η κυβέρνηση της Ρουμανίας υποστηρίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ρουμάνων ενώ η Προεδρία της Ρουμανία, της, ε, συγγνώμη, η δική σα Προεδρία γνωρεί τι τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ελπίζω ότι το έτος 2019 να είναι ένα έτος χωρίς ελεκτικό μηχανισμό για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να ενταχθούν πλήρως οι δύο χώρε αυτέ στο χώρο Σέγγεν. Σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος της κύριος Άνσιπ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ έντονη αυτή συζήτηση. Όπως γνωρίζουμε, κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας ε, θα έχουμε τον Brexit θα έχουμε ευρωεκλογέ. Και τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πι δέλτα πι. Και ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για 242 διαφορετικές προτάσεις. Λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα αυτά από κοινού μας είπε ο κύριος ε, Γιωχάνης την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι, ο πρόεδρος της ε, Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου εκεί ε, αντιλήφθηκα πως οι Ρουμάνοι υπουργοί τα παίρνουν πολύ στα σοβαρά αυτά. Αναμένω λοιπόν την επικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Κομισιόν και της Ρουμανικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και σας ευχόμαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Μουλτσουμέσκ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις των πρώην συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να ακούσω κάποιες προτάσεις, κάποιες λύσεις, μια θετική προσέγγιση, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, που σήμερα στρέφονται προς τα μας να δουν απαντήσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν, απαντήσεις ε, στα εφιστάμενα προβλήματα για διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, για διάφορες περιφέρειες και για διάφορες χώρες. Όπως ε, είπα, όταν πήρα το λόγο προηγουμένως, ε, δεν ήρθα να λογοδοτήσω για κάποια πράγματα. Ήρθα εδώ, στο Κοινοβούλιο, ως Πρωθυπουργός μιας χώρας, ως Πρωθυπουργός της Ρουμανίας για να βρούμε μαζί λύσεις που θα καταστήσουν ισχυρή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους πολίτες όλων των κρατών μελών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο για τα καλά του λόγια, για την εμπιστοσύνη που δείχνει η Κομισιόν στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ρουμανίας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και είμαι πεπισμένη ότι από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη συνένωση για τους φακέλους και τις προκλήσεις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα προβλήματα που τέθηκαν. Κυρία Στολοζάν, οι υπουργοί μας έχουν εμπειρία. Έχουν ασκήσει τη σκιώδη προεδρία και έχουν έρθει σε επαφή τόσο με τις προεδρίες των Επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με τους ε, επιτρόπους σε σχέση με τα διάφορα ζητήματα και φακέλου. Σίγουρα υποστηρίζουμε την... Ε, μας υποστηρίζει και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. ήθελα να μην θεωρήσετε ότι οι υπουργοί δεν θα χειριστούν τους φακέλους ή δεν θα μπορέσουν να δώσουν θετικές απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν επιλύσουν. Από τη δική σας πλευρά αναμένω να έχετε εμπιστοσύνη στους υπουργούς της Ρουμανίας και στην ικανότητα της Ρουμανίας. Αναφερθήκατε στην υποχρέωση της ε, Πρωθυπουργού να συναντηθεί με τους Πρωθυπουργούς της Γαλλίας ή των κατοχωρών. Είμαι ανοιχτή στο να το κάνω αυτό, είμαι ανοιχτή στο να μεταβώ στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και στο να διαβιβάσω στον πρόεδρο, τον πρόεδρο της ε, Ρουμανίας να προσεγγίσει αυτά τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί ο πρόεδρος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωζώνη, το Δεκέμβριο του 2018 ε, ορίσαμε το έτος ε, ότι θα μπούμε στο ευρώ και πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως εμείς έχουμε κρατήσει το λόγο μας και αν θέλετε το πρόγραμμα αυτό είμαστε στη διάθεσή σας να σας το παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ τον ε, πρόεδρο της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, για την υποστήριξη και του εγγυόμαστε ότι υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου. Ταυτόχρονα σεβόμαστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα όσων έχουν υποφέρει λόγω λανθασμένων αποφάσεων της δικαιοσύνης. Κύριε Φερχόφστατ, λυπάμαι ε, που έφυγε ο κύριος Φερχόφστατ από εδώ. Θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι εμείς γνωρίζουμε τους φακέλους και τις προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς γι' αυτό ζήτησα συνένεση, γιατί χρειαζόμαστε τη συναπόφαση, χρειαζόμαστε τη συνένεση και θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, περίμενα ότι ένας επικεφαλής ε, πολιτικής ομάδας ε, να κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Όχι να κάνει παρατηρήσεις για τα ιστορικά προβλήματα μιας χώρας που μόλις ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους αξιοπιστίας νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάει κανείς γνωρίζοντας ε, τα γεγονότα. Και θα ήθελα να μου πει ο κύριος Ερχόστατ σε τι έχει να επιπλήξει τη ρουμανική κυβέρνηση τις καταλογίζει και ταυτόχρονα ζητώ από τον κύριο Φερχόφστατ να αφήσει τους Ρουμάνους να αποφασίσουν μόνοι τους ε, να μην προσπαθεί να παρουσιάσει τις δικές του πεπιθήσεις ε, στους Ρουμάνους, να μην προσπαθεί να περάσει τις δικές του πεπιθήσεις στους Ρουμάνους. Είμαι πεπισμένη ότι οι συνάδελφοί μου θα παρουσιάσουν προτάσεις ε, για τις άλλες χώρες, όμως θα πρέπει να αφήσουμε τον κάθε λαό και τους πολίτες της κάθε χώρας ε, να ε, επιλέξουν ε, και να δράσουν βάσει των δικών τους πεπιθήσεων. Κυρία Κέλλερ. Είπατε ότι χιλιάδες Ρουμάνοι βγήκαν στο δρόμο για να ζητήσουν μια καλύτερη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν ε, τι σημαίνει καλή διακυβέρνηση στη Ρουμανία. Έχουμε οικονομική ανάπτυξη πάνω από 4%. Το έλλειμμά μας ε, είναι 2,96%. Ενεργεία κάτω από 4%. Οι επενδύσεις στη Ρουμανία αυξήθηκαν πάνω από 10%. Και πιστεύω αυτό σημαίνει καλή διακυβέρνηση. Και πιστεύω ότι η παραπληροφόρηση κάποιων συναδέλφων ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, οδήγησε σε αυτή την αντίληψη. Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω όλα τα αριθμητικά στοιχεία και όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση της Ρουμανίας για να διαβεβαιώσει την βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης και μια καλή διακυβέρνηση για τη Ρουμανία και τους Ρουμάνους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκρίνετε και με τα αποτελέσματα άλλων χωρών και τότε θα καταλάβετε ότι η Ρουμανία έχει μια κυβέρνηση η οποία ξέρει τι πρέπει να κάνει και η οποία έχει ασχοληθεί με τα προβλήματα των Ρουμάνων και της Ρουμανίας. Ο κύριος Πάξας ε, μας ε, ρώτησε γιατί ε, το ενδιαφέρον για την Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαταστάθηκε με τη διέρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να τη θέσουμε όλοι μας. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και να δούμε τι μας ενώνει και να δούμε και να εκτιμήσουμε λιγότερο αυτά που μας χωρίζουν. Γιατί μόνο αν είμαστε μαζί ενωμένοι, μόνο μέσω της συνοχής, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Ζωάο για τα πολύ καλά της λόγια. Πράγματι, η Σύνοδος Κορφής στο Συμπίου θα μας δώσει την ευκαιρία μαζί να χαράξουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι μίλησε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να μιλάμε συγγνώμη, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει να βρίσκουμε μαζί ανεξάρτητα της πολιτικής μας ομάδας ε, την καλύτερη δυνατή λύση που να είναι κοντά στους πολίτες έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό και το καλύτερο δυνατό μέλλον για τους πολίτες της Ένωσης. Κύριε Χόκμαρ, και η κυβέρνηση θα πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Πολλές φορές ε, το έχω πει. Δεν έχουμε κανένα νομοθέτημα επιτάπητο στο τραπέζι της κυβέρνησης που αναφέρεται στην αμνηστία. Δεν θέλουμε να υπερασπίσουμε κανένα, θέλουμε μόνο να προστατεύσουμε τους πολίτες των οποίων έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ όταν, όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, όλοι να αγωνιστούμε κατά της διαφθοράς. Και η κυβέρνηση της Ρουμανίας θα το πράξει αυτό. Όμως ε, ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν πληγεί από αποφάσεις της δικαιοσύνης, από τα μυστικά πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ της δικαιοσύνης και των μυστικών υπηρεσιών. Αυτοί που τώρα φωνάζουν δυνατά και δηλώνουν ότι αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ότι θέλουν να αγωνιστούν υπέρ του κράτους δικαίου, πολλοί από αυτούς θα κρύψουν τι συνέβη στην πραγματικότητα στη Ρουμανία. Και μάλιστα ήταν μέρος αυτού του συστήματος που οδήγησε στην ε, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Μαρινέσκου, η δική σας θέση κατά της κυβέρνησης της Ρουμανίας είναι αδικαιολόγητη. Είπατε ότι υπήρξαν επιθέσεις στην κυβέρνηση, ε, της κυβέρνησης συγγνώμη, κατά της δικαιοσύνης. Εγώ δεν θυμάμαι και κανείς ούτε ένας Ρουμανός πολίτης ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας έλαβε κάποια απόφαση κατά της δικαιοσύνης. Όλοι οι νόμοι που αναφέρονται στη δικαιοσύνη ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας και το Ρουμανικό Κοινοβούλιο εκφράζει την ψήφο των Ρουμάνων πολιτών. Μιλήσατε για ευρωπαϊκά κονδύλια, για ευρωπαϊκά ταμεία. Νομίζω ότι αναφερόσασταν στην τεχνοκρατική κυβέρνηση, γιατί εμείς κατά την ε, δική μας περίοδο διακυβέρνησης ε, μέσα σε ένα χρόνο ε, ανακτήσαμε τα ποσά, έχουμε πολύ καλή απορρόφηση των κονδυλίων για να μην μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στον τομέα της γεωργίας, Είναι του 27% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εγώ πιστεύω ότι ε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή υποστηρίζει τους πολίτες έχει αποδεικτεί από τα μέτρα που υιοθετούμε και όχι από αυτούς που ψήφισαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της ίδιας τους της χώρας. Κυρία Μπρέσο, πράγματι η εδαφική σύγκληση είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να αφήσουμε να καθυστερήσει καμία περιφέρεια. Εμείς ε, όλες τις προτάσεις σας θα τις δεκτούμε με ανοιχτό πνεύμα για να προωθήσουμε το θέμα αυτό στο θεματολογιό μας. Είπατε ότι 20 εκατομμύρια νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και τι μπορούμε να κάνουμε για να τους πείσουμε να έλθουν στις κάλπες. Καταρχήν, θα πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε λύσεις για αυτούς. Δεύτερον, θα πρέπει να δείξουμε ότι η δική μας διένεξη δεν είναι μεταξύ πολιτικών ομάδων, μεταξύ πολιτών του ίδιου κράτου μέλου, αλλά ότι οι δικές μα διαφωνίες και οι δικέ μας λύσεις είναι για αυτού. Ότι μπορούμε να αφαιρούμε προσθέμενη αξία και ότι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων που λαμβάνουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και έχω την πεποίθηση ότι μαζί μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Έχω εμπιστοσύνη στους ευρωβουλευτές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο, ότι μαζί θα μπορέσουμε το επόμενο αξάμεινο να δώσουμε τις απαντήσεις που περιμένουν αυτά τα 20 εκατομμύρια νέων, τις απαντήσεις που περιμένουν τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Γιάροκα, ελπίζω να μην ε, προφέραν σημαίνει το όνομά σας. Μας είπατε ότι είμαστε ένα φτωχό κράτος και θα, πρέπει να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο έτος ακριβώς αυτό κάναμε. Έχουμε βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης. Είδαμε ότι η λιτότητα δεν αποτελεί λύση για τη χώρα μας, ούτε και για άλλα κράτη-μέλη. αυξήσαμε τους μισθούς, αυξήσαμε τις συντάξεις, αυξήσαμε τους μισθούς των γιατρών ε, και των ε, εκπαιδευτικών Αυξήσαμε τα επιδόματα για τους ευπαθείς πληθυσμούς και ε, προσθέσαμε το περιβάλλον και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε για να μην μιλάμε για ανέχεια πέρα από τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε σχέση με την τελευταία ερώτηση, θέλω να απαντήσω στις τελευταίες κατηγορίες. Σκέφτηκα πολύ αν αξίζει ή δεν αξίζει να δώσω την απάντηση αυτή. Όμως εγώ πιστεύω ότι ως πολίτες θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ μιας εχθρικής συμπεριφοράς και μια ανοιχτή συμπεριφοράς. Κύριε Πρέντα, η κυβέρνηση της Ρουμανίας και ο πρωθυπουργός, ή πρωθυπουργός της Ρουμανίας δεν επικρίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάντοτε υποστήριξα τη φιλοευρωπαϊκή στάση μετά από 9 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου δεν δημιούργησα κανένα σκάνδαλο, όπως εσείς, δεν έκανα καμία σκηνή, ε, όπου συμφώνησα με όλες τις θετικές λύσεις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ τώρα κατά αυτών των ε, θεσμικών οργάνων. Ε, εγώ άσκησα κριτική στο ψήφισμα γιατί πίστευα και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτήν την ενότητα. Μιλήσατε για τις διαδηλώσεις ε, της 10ης Αυγούστου στη Ρουμανία. Τι λέτε για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Ποια στάση έχετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα αυτό γιατί η Γαλλία λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις. Όμως, ούτε κανένας, ούτε κάποιος Γάλλος βουλευτής, ούτε κανένας Ευρωπαίος βουλευτής ήρθε εδώ για να επικρίνει τη χώρα του, τη Γαλλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι η δική μας στάση μετρά για τους πολίτες που μας βλέπουν από το σπίτι τους κάνατε μια πολύ σοβαρή δήλωση σε σχέση με την ελευθεροτυπία. Σας διαβεβαιώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, διαβεβαιώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει παραπληροφόρηση. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Πράγματι, ένα τηλεοπτικό κανάλι είδε να διακόπτει η εκπομπή του για 10 λεπτά. Αυτό αποφασίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Η ρουμανική κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ζήτημα. Όμως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να δούμε για να δώσουμε περισσότερη αξιοπιστία στις δικές μας αποφάσεις, να είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις που κάνουμε. Και αυτά που λέμε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά όλοι μας θα κριθούμε. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα κρυθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που χρήζει ενός καλού μέλλοντος. Σας ευχαριστώ και πάλι Βασίζομαι στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην διαδρομή μας. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και τώρα η μερίσια διάταξη προβλέπει